Να περάσουμε τώρα στις επεξηγήσεις ψήφου. Πρώτη η κυρία Μαρή Κριστίν Αγνοτού. Monsieur Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι στην αίθουσα η κυρία Αρνοτή. Παρακαλώ αγαπητοί συνάδελφοι, ε, λέει ο Πρόεδρος. Παρακαλώ, φιλικά σας παρακαλώ να ε, σταματήσουν οι συζητήσεις και ενδεχομένως αν ε, θέλετε να βγείτε, αν θέλετε να συνεχίσετε τη συζήτηση σας, είναι θέμα σεβασμού προς τους ομιλητές. Η κυρία Αγνωτίου. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ψηφίσαμε κατά της επικύρωσης αυτών των συμφωνιών. Η Ουκρανία ε, αυτή τη στιγμή ε, είναι διχασμένη ανάμεσα στη Δύση και την Ανατολή και το διαπιστώνουμε καθημερινά με τραγικό τρόπο. Να μην ξεχνάμε ότι αυτή η κρίση προκύπτει, οφείλεται μάλλον ε, από στην υπογραφή ή όχι της σημερινής συμφωνίας γιατί ξεκίνησε με την αλλαγή πολιτικής του Προέδρου Γιαννούκοβιτς που μετά ανετράπη μέσω πραξικοπημάτων γιατί λοιπόν να υπογράψουμε μια τέτοια συμφωνία και να οξύνουμε την κατάσταση αντί να προσπαθήσουμε να ε, ηρεμήσουμε τα πνεύματα στις δύο πλευρές. Στόχο έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθήσει και να διατηρήσει την ειρήνη και τη σταθερότητα. Για την ώρα ε, καταλήγουμε στο ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Εν τω μεταξύ, πώς θέλετε να εφαρμόσετε μια συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών με μια χώρα στην οποία ε, μένεται φίλος πόλεμος ε, σε περίπου ένα τρίτο της επικράτειας. Ε, είναι πραγματικά ανησυχητικό και κρίμα που δεν έγινε καμιά μελέτη αξιολόγησης του αντικτύπου, διότι αυτή η συμφωνία περιέχει πολλούς κινδύνους τόσο για τους Ευρωπαίους ε, μισθωτούς και άρα τους Γάλλους μισθωτούς, αλλά όσο και για τους Ουκρανούς μισθωτούς. Σας ευχαριστώ. κύριε που έχει το λόγο είναι ο Ζαν luc Σαχοζέρ. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Καταψηφίσαμε τη συμφωνία αυτή. Μια συμφωνία σύνδεσης σήμερα σημαίνει προετοιμάζουμε τον πόλεμο. Σημαίνει ότι εντείνουμε τις εντάσεις μεταξύ Ανατολής και Δύσης, ενώ αντίθετα θα έπρεπε να δουλέψουμε υπέρ της ενότητας και της ειρήνης. Σημαίνει επίσης ότι σεβόμαστε, αν ψηφίσουμε κατά, και τον ίδιο το λαό της Ουκρανίας που έχει ψευδείς ελπίδες από την Ευρώπη, με πιο ακριβή ενέργεια, 50% πιο ακριβή, με καταστροφή θέσεων απασχόλησης, περισσότερη ενεργεία. Η Δύση δεν θα μπορέσει να ανοικοδομήσει μια διχασμένη και κατεστραμμένη χώρα. Έτσι φέρουμε ψευδεστήσεις στην Ουκρανία. Γιατί η Ουκρανία θα βρεθεί πιο φτωχή ακόμα και η Δύση δεν θα μπορέσει ποτέ να αντισταθμίσει την κατάσταση στο ύψος των προσδοκιών της Ουκρανίας, η οποία θα νιώσει προδομένη από τη Δύση τελικά. Τέλος, πρόκειται για τη δημοκρατία την ίδια στην Ουκρανία, η οποία είναι πολύ ευάλωτη και εύθραυστη. Με διαφθορά, με φασιστικά στοιχεία, τα οποία είναι υπέρ του μίσους και του ρατσισμού. Τελειώστε παρακαλώ, τέλειωσε ο χρόνος σας, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σαφόζε. Επόμενος ομιλητής, Πέτσα Γιά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ υπερψήφισα τη Συμφωνία Σύνδεσης, γιατί κατά τη γνώμη μου δεν είναι το τέλος, αλλά η αρχή μιας διαδικασίας αυτό και μέσω κοινή εργασίας και εταιρικών σχέσεων μπορούμε να την προωθήσουμε. Οποιο διαβάσει τη συμφωνία, όποιο δει τις προοπτικέ, καταλαβαίνει ότι δεν είναι θετικό μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ουκρανία, μπορεί να είναι θετικό και για την ε, Ρωσία μέσω ενός τριμερούς διαλόγου. Επαναλαμβάνω, μέσω κοινή εργασίας, μέσω εμπορίου μπορούμε να δημιουργήσουμε εμπιστοσύνη και γι' αυτό νομίζω υπερψήφισε το σώμα μας κατά πλειοψηφία αυτή τη συμφωνία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Γιάρ. Παρακαλώ τον Σάφο Λάγκενμπρουκ και άλλους να συνεχίσουν τις συζητήσεις τους εκτός εθούσης. Βέρνα, Έλμαρ, σας παρακαλώ περάστε έξω. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενη, η Κριστίνα Μόρβαε. Ευχαριστώ ως Ουγγαρέζα ε, λογικά καταψήφισε αυτή τη συμφωνία. Δεν μπορώ να ψηφίσω υπέρ μια συμφωνία ε, σύνδεσης μεταξύ Ένωσης και μιας χώρας. Ποια χώρας, τι κράτος είναι αυτό. Είναι ένα κράτος που, που καταπατεί τα ανθρώπινα δικαιώματα μιας ε, Ουγγρικής μειονότητας 200.000 ατόμων στην, στην υπερκαρπαθιακή περιοχή. Τα άτομα αυτά στην ουσία είναι υποχρεωμένα και πιέζονται να εγκαταλείψουν τη χώρα. Η συμφωνία λέει ότι η συμφωνία θα πρέπει να, ε, οι υπογράφοντες θα πρέπει να τηρούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν είναι θέμα μικροπολιτικών υπολογισμών αυτό, είναι θέμα αρχής. Όταν ε, είδα τους ε, ευρωβουλευτές από το Φιντές να υπερψηφίζουν και να χειροκροτούν πραγματικά αισθάνθηκα μεγάλη οργή ο βουλευτής από την περιοχή αυτή που εκπροσωπεί τους πολίτες αυτούς δεν μπόρεσε καν να πάρει το λόγο και αυτό με εκπλήσει ιδιαίτερα ευχαριστώ κυρία Μόρβαη ο κύριος Μάχ Ε, είναι παρόν ο κύριος Μαχ. Όχι, ωραία. Ο Νέιθεν Γκίλ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Μια συμφωνία σύνδεσης είναι κατά σε μια εμπορική συμφωνία και ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτή είναι η δεύτερη απόπειρα της Ουκρανίας για συμφωνία σύνδεσης. Η πρώτη κατέληξε σε διακοπή της δημοκρατικής διαδικασίας και στον φίλιο πόλεμο που έχουμε σήμερα στη χώρα αυτή. Ο Πούτιν συνεχίζει με την ρητορική του. Πού θα φτάσουμε όμως. Η Ουκρανία είναι μια ζώνη ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και την Ρωσία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι βγάζει αυτή την ε, ζώνη, αλλά ελπίζουμε ότι τα τάγκς του Πούτιν δεν θα καταλήξουν πιο πέρα. Λοιπόν, τι κάνουμε σήμερα. Σήμερα ρίχνουμε πετρέλαιο, ρίχνουμε βενζίνη στη φωτιά. Ο Πούτιν δεν είναι η μεγαλύτερη απειλή για τον πολιτισμό μας. Η μεγαλύτερη απειλή για τον πολιτισμό μας είναι ο μουσουλμανικός εξτρεμισμός. Αυτός, αυτό είναι το πιο επικίνδυνο και γι' αυτό ακριβώς καταψηφίσαμε τη συμφωνία αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και ευχαριστούμε που τηρήσατε το χρόνο σας. Ο καθηγητής Μπούχνερ των Πρασίνων. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, η συμφωνία λέει ε, ορισμένα πράγματα που ε, ορισμένοι δεν τα καταλαβαίνουν. Και αυτό βέβαια ε, δεν μας εκπλήσει γιατί είναι τόσο εκτεταμένο το κείμενο. Για παράδειγμα το άρθρο 89 για το εμπόριο. Εκεί λέει ότι οι νόμοι στην Ουκρανία πρέπει να τροποποιηθούν ούτω ώστε να υπάρχει προστασία των επενδύσεων και να υπάρχει δυνατότητα διαιτησίας. Προστασία των επενδύσεων. Τι σημαίνει αυτό. Ότι η Ουκρανία δεν θα πρέπει να εισαγάγει νέους κοινωνικούς και ε, επενδυτικούς νόμους που μειώνουν τις δυνατότητες κέρδους από τους Ευρωπαίους επενδυτές. Αυτό μειώνει τη δημοκρατία και όπως ξέρετε οι διαδικασίες διαιτησίας μπορεί να οδηγήσουν σε πρόστιμα δισεκατομμυρίων που θα κατέστρεφαν την Ουκρανική βιομηχανία ή τουλάχιστον θα τις έκαναν μεγάλες ζημιές. Αν ε, λοιπόν υπογράψουμε μια τέτοια συμφωνία ο λαός της Ουκρανίας πολύ σύντομα θα διαπιστώσει ότι έχουμε αποστείλει δούριο ύπο στην Ουκρανία. Θα χαθεί εμπιστοσύνη στην Ευρώπη, οι σχέσεις μας θα υποστούν μεγάλη βλάβη. Επαναλαμβάνω, μια συμφωνία με την Ουκρανία είναι απόλυτα απαραίτητη. Αλλά παρακαλώ όχι με τέτοια μορφή, όχι με τέτοιε ρήτρε. Ευχαριστώ πολύ καθηγητά Μπούχνερ. Επόμενη η Τατιάνα Ζδάνοκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταψήφισα την συμφωνία αυτή. Πιστεύω ότι δεν έχει προετοιμαστεί καλά, ότι είναι ανεύθυνο. Είναι μια ιδιαίτερα πολιτική απόφαση. Σε τρεις μέρες έχουμε μια σημαντική επέτειο, 51 χρόνια θα έχουν περάσει από μια αντίστοιχη συμφωνία που κάναμε με την Τουρκία. Και πού βρίσκεται σήμερα η σχέση μας ε, με την Τουρκία. Συστήνω λοιπόν να το θυμίζουμε αυτό σε αυτούς τους αφελείς ε, ονειροπόλους στην Ουκρανία που ελπίζουν ότι πολύ γρήγορα θα ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ή ότι θα έχουν ε, κατάργηση των θεωρήσεων είναι ανέθυνο να υπόσχεται τέτοια πράγματα στους Ουκρανούς ο κύριος Ποροσέγκο. Συνεπώς ζητούμε από τους νέους εδώ να ξέρουν ότι είναι μια χώρα Ουκρανία η οποία πρέπει να ανοικοδομηθεί και ότι η απόφασή μας αυτή είναι εντελώ ανεύθυνη. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Σντάνακα. Επόμενος ομιλητής, η κυρία Γκίλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υπερψήφισα εγώ την έκθεση Σάριου Βόλσκι, γιατί πιστεύω ότι η ενίσχυση των δεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ουκρανία σε αυτό το στάδιο που βρισκόμαστε είναι ζωτική σημασία. Η Ουκρανία είναι μια γείτονα χώρα η οποία έχει σταθερότητα και η σταθερότητα αυτή επηρεάζει πολύ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ότι είναι προς το συμφέρον των πολιτών εκατέρωθεν να δεσμευτούμε υπέρ της Ουκρανίας και να τη στηρίξουμε στις προσπάθειές της για μεταρρυθμίσεις, για οικονομικές και πολιτικές αλλαγές. Με στενή συνεργασία επίσης στο θέμα της ασφάλειας στην περιοχή. Πιστεύω επίσης ότι η συμφωνία αυτή βοηθάει για να καταλήξουμε σε μια πολιτική λύση όσον αφορά την κρίση της σημερινής στην Ουκρανία και όσον αφορά την εδαφική κυριαρχία, εδαφική μαλακερότητα και κυριαρχία στην Ουκρανία. Υπάρχει και η συμφωνία της EFT ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την, ε, ε, και την Ουκρανία. Καθυστερούν τα πράγματα εξαιτία της κρίσης εκεί. Όμως ένα τέτοιο βήμα μπορεί να είναι αναγκαίο για να αποκλιμακωθεί η κατάσταση. Όμως θέλω επίσης να πω ότι η απόφαση της Ουκρανίας να επικυρώσει την συμφωνία αυτή σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση προέρχεται από ένα κυρίαρχο κράτος και εμείς το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να στηρίξουμε τις επιλογές μιας κυρίαρχης χώρας. Πρόεδρος, οι επεξηγήσει ψήφου περιορίζονται σε ένα λεπτό. Θέλω να επιθυμίσω στους συναδέλφους Παρακαλώ να τηρείτε το χρόνο σας. Πίτρο Μαχ, ο οποίος βλέπω ότι έχει επανέλθει. Έχετε το λόγο. Σα ευχαριστώ κυρίες και κύριοι. Εγώ καταψήφισα τη συμφωνία αυτή γιατί πιστεύω πως δεν είναι προς όφελος της Ουκρανίας κυρίως. Είμαι υπέρ του ελεύθερων συναλλαγών. Όμως η Ουκρανία δεσμεύτηκε να υιοθετήσει το σύνολο του κεκτημένου, όλους τους κανονισμούς και τις οδηγίες της Ένωσης. Αυτή η συμφωνία δίχασε πολιτικά την Ουκρανία τον Νοέμβριο, οδήγησε στη ε, Μαϊντάν ήταν ε, προς όφελος της δυτικής χώρας, δηλαδή η Τελωνιακή Ένωση με την ε, Ένωση ήταν πλονεκτική για την ανατολική, το ανατολικό κομμάτι της χώρας, ενώ όχι με το, για το δυτικό, που, γιατί καθιστά πιο δύσκολο το εμπόριο με την ε, Σοβιετική Ένωση, λέει ο μιλητής είναι βάρος η υιοθέτηση του συνόλου του κεκτημένου για τις στοχές χώρες της Ένωσης και σίγουρα θα είναι και για την Ουκρανία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που επίσης για ακριβώς ένα λεπτό. Τόμας Ζεχόφσκι. Είναι επεξήγηση ψήφου για την ε, έκθεση Μωράης και μετά είναι η κυρία Κοράτσα και με αυτό κλείνουμε τις επεξήγησεις ψήφου. Ο κύριος Ντεχόφσκι. Ευχαριστώ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για το που μου δώσατε το λόγο. Εγώ υπερψήφισα αυτή την έκθεση γιατί πιστεύω πως ε, είναι ένα μικρό βήμα για την Ένωση και για την Ουκρανία, αλλά είναι ένα τεράστιο βήμα για όλους μας ε, προς όφελος της ειρήνης και της ε, σταθερότητας στην Ουκρανία. Ξέρω ότι περάσαμε εμείς ως ε, Τσέχοι όταν παρόμοια συμφωνία υιοθετήθηκε. Θυμάμαι τις συζητήσεις που έγιναν τότε στην, στα παλαιά κράτη-μέλη της Ένωσης για το ότι αυτή η συμφωνία θα έτσι σε κίνδυνο την σταθερότητα ή ότι θα είχε αρνητικές επιπτώσεις για τα νέα μέλη. Ωστόσο, αυτό δεν επαληθεύθηκε και ελπίζω πως το ίδιο θα συμβεί και τώρα για την Ουκρανία. Και ότι αντιθέτως η συμφωνία αυτή θα καταστήσει την Ευρώπη και την Ουκρανία πιο ευημερούσες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε. Τελευταία ομιλήτρια για τις επεξηγήσεις ψήφου η Άννα Μαρία Κοράτσα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τη στιγμή που ο κύριος Πούτεν ε, δοκιμάζει τις ε, αδυναμίες μας και προσπαθεί να εκφοβήσει με στρατιωτική δύναμη που ο κορονικός λαός είναι αντικείμενο εισβολής, ε, είναι σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να είναι ενωμένο με μεγάλη πλειοψηφία ώστε να δείξει τη στήριξή του. Εγώ υπερψήφισα τη Συμφωνία Σύνδεσης με την Ουκρανία με όλη μου την καρδιά. Είναι πάρα πολύ σημαντική οικονομικά, αλλά είναι και πολύ, ένα σημαντικό πολιτικό μήνυμα να μην δεχτούμε αυτού του είδους τις ενέργειες, αυτού του είδους ε, τη συμπεριφορά στην Ευρώπη. Αγωνίζονται για την ελευθερία, την επικυριαρχία τους, την ε, ακεραιότητα της, ε, την εδαφική τους είναι πολύ σημαντικό ότι η άκρα δεξιά και η άκρα αριστερά καταψήφισαν αυτήν τη συμφωνία είναι απαράδεκτο και είναι εκτός των ευρωπαϊκών αξιών τις οποίες όλες στηρίζουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι κλείνουν οι επεξηγήσεις ψήφου. Διακόπτεται η συνεδρίαση μέχρι τις 3 το απόγευμα.